Λοιπόν, τώρα κάποια σχόλια. Στην αρχή της ε, συνεδριάσεώς μας θα ήθελα να καλωσορίσω τη Μαρία Ρωμάνα Ντεκάσπαρη, τη θυγατέρα του μεγάλου ηγέτου Αλτσίντε Ντεκάσπαρη, που ήταν ένας από τους ιδρυτές πατέρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης.